Οπότε δίνω συγχρονισμό τον λόγο στην κυρία Ντιρόν για δύο λεπτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, την παραμονή της ε, πεντηκονταετίας από την ανεξαρτησία του Κονγκό, μας φαίνεται σημαντικό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να αποφανθεί για τη δολοφονία του κ. Σεμπάγια. Ο κ. Σεμπάγια είναι ένας υπερασπιστής των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, είναι πρόεδρο τη μη κυβερνητική οργάνωση Η Φωνή των Μη Εχόντων Φωνή. Βρέθηκε δολοφονημένο ε, στο αυτοκίνητο του στι 2 Ιουνίου ε, του 2010 στην Κινσάσα και ε, αγνοείται και η τύχη του οδηγού του. Τα ερωτήματά μου είναι τα εξή. Για ποιο λόγο δολοφονήθηκε, από ποιον. Όπω λέει και το ψήφισμα, νομίζω ότι μια ανεξάρτητη αξιόπιστη και διαφανής ε, έρευνα πρέπει να γίνει για να διαβριθούν τα αίτια του θανάτου του κ. Σεμπάγια και για να δούμε γιατί έχει εξαφανιστεί ο οδηγός του. Ξέρουμε ότι υπάρχει γενικά κατάπτωση των ε, ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Κονγκό και αυτό μας ενισχύει πάρα πολύ. Πάρα πολλοί περασπιστές ε, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, διάφοροι δημοσιογράφοι, ε, ακτιβιστές ε, έχουν εξαφανιστεί, δεν ξέρουμε γιατί. Οι έρευνες από τις στρατιωτικές αρχές ε, γίνονται, αλλά με τρομερές παρατυπίες. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να δούμε ποιοι είναι οι υπεύθυνοι της δολοφονίας, να διωχθούν, να παραπαινθούν στη δικαιοσύνη και θα πρέπει να συσταθεί μια ερευνητική επιτροπή διεθνούς εμβέλειας για να τιμωρηθούν οι ένοχοι. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό για τη δημοκρατία, το υπενθύμισαμε και σήμερα το πρωί στην, στα πλαίσια της έκθεσης Χάουταλα. Η Συμφωνία του Κοτονού μιλάει για το σεβασμό των ανθρωπινών δικαιωμάτων. Γι' αυτό ακριβώ μέσω του ψηφίσματο ζητάμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση καθώ και από τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονκό να στρέψουν τα την προσοχή τους προς αυτό το θέμα. Το Κοινοβούλιο θα πρέπει να ζητήσει από τις κονγκολέζικες αρχές να συμμορφωθούν με τη δήλωση για τα ανθρώπινα δικαιώματα που υιοθέτησαν το 1998 ε, στη συνέλευση ε, του ΟΗΕ και όλα τα μέτρα που σκοπεύουν να προστατεύσουν τους ακτιβιστές και υπερασπιστές των ανθρωπινών δικαιωμάτων. Αυτό το μήνυμα θα στείλω στην Κινσάσα όταν εορταστεί η 50η επέτειος από την εξαρτησία στην 30η, την 30η Ιουνίου του 2010. Ευχαριστώ. κύριος Κατσμάρα και ένα λεπτό. Κυρίες και κύριοι, χτες μιλήσαμε για την προστασία των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων γενικότερα. Σήμερα έχουμε μια ειδική περίπτωση, μια πολύ συγκεκριμένη περίπτωση, αυτήν του κυρίου Τσεμπέγια ε, ο οποίος ήταν υπερασπιστής των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ε, από ό,τι φαίνεται δολοφονήθηκε εξαιτία τη δράση του. Οι δράστες προφανώ είχαν τα δικά του κίνητρα, τα οποία γνωρούμε αυτή τη στιγμή. Όμω γνωρίζουμε ένα πράγμα. Οι στόχοι των δραστών ήταν αντίθετοι με του δικού μα στόχου, που είναι η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Οι υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων καταδιώκονται και διώκονται διότι ε, βελτιώνουν τη συνειδητοποίηση εκ μέρους της κοινής Και θα πρέπει οι δράστες να συλληφθούν, να τιμωρηθούν και να εξηγηθεί αυτό το έγκλημα. Να διαλευκανθεί. Η έρευνα θα πρέπει να είναι ανεξάρτητη και αυτό ζητούμε στο ψήφισμα μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ για ένα μισή λεπτό η κυρία Βερζιά. Euh, Η δολοφονία του Φλωριμπέρ Σεμπάγια Μπενζίρε ε, διευθυντή της οργάνωσης ε, η φωνή αυτών που δεν έχουν φωνή τη στιγμή που τον είχαν συγκαλέσει στην αστυνομία καθώς και εξαφάνιση του οδηγού του είναι συμβολική σημασία για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Κονγκό. Διερωτώμαστε γιατί η οικογένεια του κ. Σεμπάγια δεν μπορεί καν να έχει πρόσβαση στο πτώμα του. Ο κ. Σεμπάγια ήταν γνωστό για τι θέσει που είχε υπερασπιστεί εναντίον των Κογκολέζων ηθινών, κατήγγειλε συστηματικά στα ΜΜΕ, στις μη κυβερνητικέ οργανώσεις, τη δραματική κατάσταση στο Κονγκό. Ε, είναι αναρρύθμιτοι οι υπερασπιστές ανθρωπινών δικαιωμάτων, οι δημοσιογράφοι που απειλούνται, βασανίζονται και σκοτώνται σε αυτή τη χώρα. Το 2005 ένας άλλος ε, υπερασπιστής ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ο κ. Σενκίχε και η γυναίκα του ο Σέρας Μασέη το 2007, το 2008, άλλοι υπερασπιστές. Είναι λίγα παραδείγματα μέσα στα πολυάριθμα θύματα. Τη στιγμή που το Διεθνές, Δικαστήριο της, το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο εξέδιδε ένα ένταλμα σύλληψης εναντίον διαφόρων ηθινόντων, τη στιγμή που η κατάσταση οικονομική και κοινωνική στη χώρα επιδεινώνεται, τη στιγμή που το κλίμα είναι πάρα πολύ άσχημο στη χώρα. Έχουμε δολοφονίες, έχουμε στρατολογήσεις παιδιών στρατιωτών. Η κατάσταση είναι αποτρόπαια. Επίσης υπάρχει μια συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση, Συμφωνία Κοτονού. Στα πλαίσια αυτά, ε, οι κογκολέζικες αρχές ε, δεσμεύτηκαν να σεβαστούν τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αν δεν κάνω λάθος, Πρόεδρε, ζητώ συγγνώμη. Έχω δύο Σας ευχαριστώ, αγαπητοί συνάδελφοι. Ενάμιση λεπτό είχατε. 1,5 λεπτό. Σας άφησα να μιλήσετε ένα και 45 και δεν είναι η πρώτη φορά. Ε, σας παρακαλώ. Δεν πρέπει να μιλάτε εις βάρος των άλλων συναδέλφων. Δεν, δεν γίνεται έτσι. Η κυρία Σάκε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Μιλώ ως ε, συνσυντάκτης ε, του ψηφίσματος. Το Νοέμβριο, μετά από μερικούς μήνες, η αντιπροσωπεία του Κοινοβουλίου μας θα βρεθεί στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. όπου θα συνεδριάσει η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ευρωπαϊκής Ένωσης χωρών ΑΚΕ. Θα πρέπει να καθορίσουμε τη στάση μας λοιπόν. Ποια θα είναι η στάση μας όταν κοιτάμε τα πρόσωπα αυτών που θα μας φιλοξενούν. Δεν μπορούμε να μείνουμε σιωπηλοί και μουγγί μπροστά σε αυτή την προσβολή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η πρόσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων δεν μπορεί να είναι απλώς μια κουβέντα γιατί κάποιοι πληρώνουν με τη ζωή τους βαρύ το τίμημα της προάσπισης αυτής. Θα πρέπει να ορθωθεί η φωνή μας και να ακουστεί. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Τσαρνέτσχη. Με συγχωρείτε δεν Τώρα είναι η κυρία Σάκη για δύο λεπτά. Δεν είναι εδώ η κυρία Σάκη. Οπότε τελείωσαν οι συντάκτες και περνάμε στις ομάδες. Ο κύριος Πόσελτ για ένα λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, η φρικτή τύχη του κυρίου Σύρε δεν είναι μεμονωμένη περίπτωση. Είναι η κορυφή του παγόβουνου όχι μόνο για τη Δημοκρατία του Κονγκό αλλά συνολικά για την Αφρική. Είναι μια, το Κονγκό είναι μια συναρπαστική χώρα, θα μπορούσε να γίνει πλούσια από το υπέδαφος και από την ενέργεια που έχει, η οποία θα μπορούσε να παρέχει ενέργεια σε ολόκληρη την Αφρική. Αλλά δυστυχώς συμβαίνει το αντίθετο. Το Κονγκό είναι ένας τεράστιος παράγοντας αποσταθεροποίησης που εξάγεται σε άλλες χώρες γειτονικέ. Γι' αυτό ως Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει ως βασικό σημείο της πολιτικής μας, της ειρήνευσης και της ανάπτυξης να έχουμε το Κονγκό γιατί εκεί πέρα κρίνεται η τύχη της Αφρικής. Και είναι σωστό νομίζω το ότι η επόμενη μεγάλη διάσκεψη μας λαμβάνει χώρα εκεί. Ευχαριστώ κύριε Πόσελτ, η κυρία Κρετού κατόπιν. Ευχαριστώ και εγώ θα ήθελα να καταδικάσω το έγκλημα αυτό εις βάρος ενός από τους πιο σεβαστούς αγωνιστές ε, για τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Το όνομα της ε, ΜΚΟ νομίζω ε, τα λέει όλα. Η φωνή αυτών που δεν έχουν φωνή αφιέρωσε τη ζωή του σε αυτούς τους ανθρώπους, τον παρενοχλούσαν ε, γιατί ανέφερε την διαφθορά στο στρατό και βεβαίως είδαμε πως είχε βίαιο και βάρβαρο θάνατο και αυτό λέει πολλά για τα ανθρώπινα δικαιώματα στο Κονγκό όπου έχουμε βασανιστήρια, αυθαίρετες συλλήψεις, ε, σεξουαλική βία και εκτελέσεις. Η ευρωπαϊκή διπλωματία λοιπόν θα πρέπει να επιμείνει έτσι ώστε οι αρχές του Κονγκό να ξεκινήσουν μία διάφανη και αξιόπιστη έρευνα. Πρέπει να παλέψουμε κατά της ατιμορρησίας αυτή σε μία χώρα στην οποία ο εμφύλιος πόλεμος οδηγεί σε σφαγές και βιασμούς. Νομίζω πως η αποστολή του ΟΗΕ εκεί πέρα μπορεί να βοηθήσει την έρευνα. Ευχαριστώ για ένα λεπτό ο κύριος Κόβαλ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αυτό που αντιμετωπίζουμε σήμερα, όταν η Αφρική ζητάει την υποστήριξή μας ή την συνεργασία μας, εμείς προσπαθούμε να την υποστηρίξουμε, προσπαθούμε να τη βοηθήσουμε. Υπάρχουν κάποια πρότυπα για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Υπάρχουν ε, κάποιοι κανόνες για τη διερεύνηση των ε, εγκλημάτων και θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να σεβαστεί αυτούς τους κανόνες. Το κλειδί όλης αυτής της υπόθεσης είναι το τμήμα του ψηφίσματος που μιλάει για τη διενέργεια μιας ε, εξεταστικής επιτροπής για να διερευνηθεί αυτό το έγκλημα. Ευχαριστώ. Ακολουθούν οι υπόλοιποι ομιλητέ για ένα λεπτό, κύριο Σκέλαμ. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Δυστυχώ, αυτή η δολοφονία του κυρίου Μπαχαζίρε που έλαβε χώρα πριν από 15 μέρες δεν είναι ένα μεμονωμένο γεγονό μια μεμονωμένη τραγωδία. Όπω είπε, και ο ειδικό συγητής, η ε, υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις ε, ε, συμμετοχής του κράτους. Τέτοιου είδους πολιτικές δολοφονίες αποτελούν τμήμα μιας γενικότερης τάσης παρενόχλησης και δολοφονιών, προασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δημοσιογράφων κλπ. Τα τελευταία πέντε χρόνια στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κόγκο εκφράζουμε τη βαθιά μας λύπη και συμπάσχουμε με την ε, οικογένεια του κυρίου Μπαχαζήρα και καλούμε τον πρόξενο και την ε, Κομισιόν να πιέσουν τις ε, κρατικές αρχές της δημοκρατίας, της λαϊκής δημοκρατίας του Κονγκό προκειμένου αυτές να εξασφαλίσουν κανονικές συνθήκες για την έρευνα που θα γίνει προκειμένου οι δράστες να δικαστούν. Ευχαριστώ. Για ένα λεπτά η κυρία Κόρολα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σωστό είναι να ασχοληθούμε με αυτό το ζήτημα στην Ολομέλεια. Ο άνθρωπος αυτός ήταν ένας γενναίος υπερασπιστής των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας στο Κονγκό και υπέστη διώξεις από τις αρχές. Δεν μπορέσαμε να τον προστατεύσουμε. Η δολοφονία αυτού του ανθρώπου και άλλων σέγγευτών είναι ένα φαινόμενο με αυξανόμενη συχνότητα στο Κονγκό. Τα τελευταία πέντε χρόνια σκοτώθηκαν πολλοί υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αλλά πρέπει να τονίσουμε πως ε, το σημαντικό είναι πως πρέπει να υπάρξει αυτό διάθεση και να μπορέσουν οι άνθρωποι του Κονγκό να αποφασίσουν μόνοι τους την μοίρα τους και να καταπολεμηθεί η διαφθορά και ο στρατός και η αστυνομία να ελεγχθούν. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ για ένα λεπτό ο κύριος Πρέντα. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να εκφράσω τα συλληπιτήριά μου προς την οικογένεια του Φλόριμπέρ Σεμπέγια Μπαχιζήρα. Ο θάνατός του είναι ένα τραγικό γεγονός. Ε, ήταν ένας αξιοσέβαστος υπερασπιστής ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ο θάνατός του είναι απαράδεκτος και θα πρέπει να τύχει γενικής καταδίκης, όπως είπαν οι συναδελφοί μου. Νομίζω ότι πρέπει να υπάρχει μια αξιόπιστη και διαφανής έρευνα, ούτως ώστε να διερευνηθούν τα αίτια της ε, δολοφονίας και το πώς ε, έλαβε χώρα και θα πρέπει να εμπλακεί και ο ΙΕ, ο εισηγητής ε, του ΟΗΕ ε, που ασχολείται με εξοδικαστικές δολοφονίες ε, είπε λοιπόν ότι μάλλον εμπλέκεται και το επίσημο κράτος στη δολοφονία αυτή. Αυτή η δολοφονία δείχνει μια αυξανόμενη ανησυχητική τάση στη λαϊκή δημοκρατία του Κονγκό τα τελευταία χρόνια γιατί στο Κονγκό έχουν υπάρξει πολλές δολοφονίες δημοσιογράφων, υπερασπιστών ανθρωπίνων δικαιωμάτων ε, και οι αρχές δεν κάνουν τίποτε. Ε, οι αρχές θα πρέπει να καταδικάσουν την δημορισία. Θα πρέπει να κάνουν κάτι γι' αυτό. Ευχαριστώ κύριε Πρέντα. Περνάμε τώρα σε διαδικασία και έτσι διάει. Κύριε Στάιλο για ένα λεπτό. Thank you, uh, Mr. President. I'd like to thank... Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συντάκτες του ψηφίσματος αυτού η δολοφονία του κ. Μπαχιζήρε οδήγησαν 15 οργανώσεις και τον κ. Μπάνκι Μουν τον ίδιο να ζητήσουν ανεξάρτητη έρευνα. Είχε λάβει επανειλημμένως απειλές από την αστυνομία και από ό,τι κατάλαβα την 1η Ιουνίου πριν δολοφονηθεί είχε κληθεί σε αστυνομικό τμήμα. Το πτώμα του βρέθηκε την επόμενη ακριβώς η Κομισιόν και το Συμβούλιο θα πρέπει να πιέσουν προκειμένου να γίνει μια ανεξάρτητη διερεύνηση των γεγονότων. Και θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι και η οικογένειά του θα τηρηθεί ενήμερη. Εμείς θεωρούμε ως δεδομένο, αλλά αυτός ο άνθρωπος ήταν, τα προασπιζόταν στη χώρα του και αξίζει του σεβασμού μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Κύριε Στάιλερ. Εδώ πέρα τελειώνει η διαδικασία KHDI με τον κύριο Τάνοκ. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, θυμόμαστε έτσι την ε, περίπτωση του Μομπούτου Σεσεσέκο, του γνωστού κλεπτοκράτη, στη χώρα που, που λεγόταν ε, Ζαΐρ και έγινε λαϊκή δημοκρατία του Κονγκού και οι δημοσιογράφοι απειλούνται και εκτελούνται. Το δε όνομα του Φλωριμπέρτ Τσεμπέγια Μπαζίρε είναι το τελευταίο σε μια σειρά υπερασπιστών ε, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που κλήρωσαν το υπέρτατο τίμημα για τις πεπιθέσεις τους. Θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να ενισχύσει τις προσπάθειές της ε, για να βελτιώσει την κατάσταση λαϊκή δημοκρατία του Κονγκό και η κατάσταση αυτή συνδέεται με τον έλεγχο των πόρων, ειδικά των ορυκτών. Θα πρέπει λοιπόν να ενισχυθεί η διαδικασία πιστοποίησης πέρα από τα διαμάντια και σε άλλα ορυκτά για να σταματήσει αυτή η ανομία που έχει ως αποτέλεσμα το θάνατο γενναίων ανθρώπων όπως ο κύριος Μπαχιζήρε. Ευχαριστώ κύριε Τάνοκ. Τον λόγο τώρα έχει ο κύριος πίτροπος, ο κύριος Ντελή. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί βουλευτές, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έμαθε για το θάνατο του κυρίου Μπαχίρε, Μπαχιζίρε με μεγάλη θλίψη. Ήταν ένας από τους πολύ γνωστούς υπερασπιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Ήταν επικεφαλής της οργάνωσης and Wife φωνή αυτό που δεν έχουν φωνή με την οποία συνεργαζόμαστε και είναι μία από τις πιο γνωστές και αξιοσέβαστες ε, μη κυβερνητικές οργανώσεις. Οι συνθήκες του θανάτου του ε, υποδηλώνουν ότι μάλλον πρόκειται περί δολοφονίας και μπορεί να εμπλέκονται και αξιωματούχοι του κράτους. Ο θάνατος του κυρίου Μπαχιζίρε οδήγησε σε έντονες αντιδράσεις όχι μόνο εντός του Κονγκό, αλλά και γενικά στη διεθνή κοινότητα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και διάφορα επιμέρους κράτη-μέλη, αλλά και ο ΙΕ, καθώς και οι Ηνωμένες Πολιτείες, Όλοι εξέφρασαν τις ανησυχίες τους και ζήτησαν να γίνουν σοβαρές έρευνες, ούτως ώστε να βρεθούν οι ένοχοι και να αποφευθεί η ατιμορρησία. Θα πρέπει τα γεγονότα να διερευνηθούν και οι δράστες θα πρέπει να διωχθούν. Ο πρόεδρος Καμπίλα εξέφρασε την επιθυμία του να διερευνηθούν τα αίτια του θανάτου. Κάποιοι ύποπτοι από την επίσημη εθνική αστυνομία έχουν συλληφθεί και ο επικεφαλής αστυνομίας έχει τεθεί σε διαθεσιμότητα μέχρι νεοτέρας. Οι αρχέ του Κονγκό ε, δέχτηκαν να συνεργαστούν πλήρως. Μία ε, ιατρική ομάδα θα εξετάσει το πτώμα του κυρίου Σεμπέγια Μπαχιζίδα και τις επόμενες εβδομάδες θα ε, ετοιμάσει ένα πόρισμα για τα αίτια του θανάτου του. Οι αρχές καταλαβαίνουν την ανάγκη να προωθήσουν μια αξιόπιστη και διαφανή έρευνα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα παρακολουθήσει εκ του σύνεγγης εξελίξεις μαζί με τα κράτη-μέλη ε, και επιτόπου στην Κινσάσα. Ενθαρρύνουν τις αρχές να προβούν σε γρήγορα αποτελέσματα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, ζητάει από την κυβέρνηση του Κονγκό να καταπολεμήσει την ατιμορρησία και θα βοηθήσει όσο μπορεί τις αρχές για να προασπίσουν τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και να σεβαστούν το κράτος δικαίου. Ευχαριστούμε κύριε Επίτροπε. Τελείωσε η συζήτηση. Έχουν κατατεθεί έξι προτάσεις ψηφίσματος από τους σοσιαλδημοκράτες, πράσινους, το ΕΛΚ, από την Ευρωπαϊκή Ρωμανία Αριστερά, τους Ευρωπαίους Συντηρητικούς και Ζωσπάστες και τους φιλελεύθερους. Η ψηφοφορία θα γίνει στο τέλος των συζητήσεων. Ακολουθεί το θέμα του Νεπάλ. Θα ζητήσω πρώτα απ' όλα από τους ε, συντάκτες να λάβουν τον λόγο και πρώτα απ' όλα η κυρία Γκέριγκερντε Ντε ε, Ευχαριστώ